που ελπίζω ότι θα μας βοηθήσει να προωθήσουμε ακόμη περισσότερο την Ένωση της Ευρώπης και να προωθήσουμε και την ειρήνη ανά τον κόσμο. Επ' αυτού του θέματος θα ήθελα τώρα να προβώ σε δήλωση. Κυρίε και κύριοι, η διάσκεψη των Προέδρων με παρακάλεσε να κάνω δήλωση για τα συμβαίνοντα στην Μέση Ανατολή. Η σχετική συζήτηση θα γίνει την Τετάρτη το απόγευμα και μάλιστα εν παρουσία του προεδρεύοντος των ε, ε, Υπουργών Εξωτερικών Τσέχου Υπουργού κ. Σφάρτσενμπεργκ. Το επισημαίνω αυτό διότι δεν ήταν βέβαιο αν θα μπορεί να προσέλθει αλλά επιμείναμε και επιτύχαμε να υποσχεθεί να προσέλθει διότι φεύγει και για την Νότιο Αφρική την ίδια μέρα θα έρθει, έστω και αν δεν θα μπορέσει να μείνει για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Κυρίες και κύριοι, ενώ στην αρχή εδώ του έτους 2009 εμείς συνερχόμεθα σε περίοδο συνόδου, εξακολουθούν να θνίσκουν άνθρωποι στην Μέση Ανατολή. Προσωπικά και νομίζω ότι οι περισσότεροι θα συμφωνήσετε, κατά την παρακολούθηση των γεγονότων αυτών στην τηλεόραση έχω έντονα το αίσθημα ότι είναι πράγματα τα οποία έχουμε ξαναδεί. Ε, στο όνομα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επιθυμώ να εκφράσω την βαθιτά τη λύπη μου για την κλιμάκωση των συγκρούσεων μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στη λωρίδα της Γάζας. Λέω με κάθε σαφήνεια ότι δεν είναι αποδεκτό να συνεχίσουν τα πάθη των ανθρώπων αυτών εκεί, να συνεχίζεται η άσκηση βίας και ταυτόχρονα μάλιστα να βάλλονται και συνεργάτες των Ηνωμένων Μέχρι πού πλέον πρέπει να κλιμακωθεί η βία μέχρι ότου μπορέσει πια να κυριαρχήσει η λογική. Πρέπει να καταπαύσουν οι βιοπραγίες και από τις δύο πλευρές. Είναι απολύτως απαράδεκτο και οφείλουμε όλοι να το καταδικάσουμε οξύτατα όταν η Χαμάς εκτοξεύει πυράβλους κατά Ισραηλινών πόλεων. Και ούτε πρέπει να λησμονούμε ότι η Χαμάς ήταν εκείνη η οποία διέκοψε την κατάπαυση του πυρός. Όμως και σε ό,τι αφορά την αντίδραση, αυτή δεν πρέπει να είναι δυσανάλογη. Όλοι οι άνθρωποι στην Μέση Ανατολή χαίρουν της ίδιας ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Η προστασία του κράτους δεν μπορεί να δικαιολογήσει κάθε είδους χρήση βίας από την οποία πλήττεται κατά πρώτον βαθμό ο άμαχος πληθυσμός. Πρέπει να προσφερθεί βοήθεια στους ανθρώπους. Η αξιοπρέπεια του Παλαιστινίου είναι ίδια όπως του Ισραηλινού ή του Ευρωπαίου ή του Αμερικανού. Όλοι οι άνθρωποι στον πλανήτη είναι ίσοι. Δεν επιτρέπεται να αποδεχθούμε οποιαδήποτε επιδείνωση της ανθρωπιστικής κατάστασης. Ως πολιτικός υπεύθυνοι πρέπει να είμαστε διατεθειμένοι και έτοιμοι να συμβάλλουμε αποφασιστικά ώστε να υπάρξει και διαρκής διέξοδος από την κλιμάκωση αυτή της βίας η μείωση του, της έννοιας της ασφάλειας σε καθαρά στρατιωτικά μόνο ε, σε στρατιωτικούς μόνο όρους δεν μπορεί να επαρκεί. Πρέπει να υπάρξει επιτέλους μια πολιτική λύση στο Μεσανατολικό. Και αυτό σημαίνει κυρίως ότι πρέπει να εξαχθούν τα απαραίτητα διδάγματα από τις αποτυχίες των μέχρι τώρα προσπαθειών. Και πρέπει οι νέες προσπάθειες να είναι προπάντων διαρκής τηλεφώνησα συχνά στον πρόεδρο του Ισραήλ κύριο Σιμών Πέρες, τον Σαλάμ Φαγιάτ, την πρόεδρο της Κνεσέτα Λιαϊτσίκ και βεβαίως και με τον ύπατο εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για εξωτερική ε, πολιτική και πολιτική ασφάλεια τον Χαβιέρ Σολάνα, ο οποίος ε, πέρασε πάρα πολλές μέρες στην περιοχή αυτή. Μίλησα και με τον αντιπρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Συνελεύσεως της Ευρωμεσογειακής Συνεργασίας γιατί έχω και την Προεδρία της Ευρωμεσογειακής Συνεργασίας αυτή τη στιγμή και με, μίλησα και με τον Ιορδανό ε, Πρόεδρο του Κοινοβουλίου και με τον Τζανφράν Κοφίνη με τον Πρόεδρο του Μαροκινού Κοινοβουλίου Μουσταφά Μανσουρί. Σε όλες αυτές τις τηλεφωνικές μου συνομιλίες κατέστησα σαφές ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστηρίζει απολύτως τις αξιώσεις που διατύπωσε το Συμβούλιο Υπουργών εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και αυτές που περιλαμβάνονται στο ψήφισμα των ΗΕ της 8 Ιανουαρίου. Είναι καταθλιπτικό κυρίε και κύριοι ότι αυτή, αυτό το νομικά δεσμευτικό ψήφισμα ενώ του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ όπου απέσχουν οι Αμερικανοί και με τον τρόπο αυτό, με την αποχή του, δηλαδή κατέστησαν δυνατόν να ψηφιστεί το ψήφισμα. Πρόκειται λοιπόν για νομικά δεσμευτικό κείμενο και όμω περιφρονείται και καταπατείται και από τι δύο πλευρέ και το Ισραήλ και την Χαμά. Κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, πρέπει να υπάρξει άμεση εκεχηρία. Η άμεση αυτή εκεχηρία πρέπει να επιτευχθεί με την διαμεσολάβηση της Αιγύπτου και με συμμετοχή όλων των μερών. Να ανοίξουν αμέσως οδοί για την διέλευση της ανθρωπιστικής βοήθειας και ο οργανισμός ε, UNRWA των Ηνωμένων Εθνών να μπορέσει να δραστηριοποιηθεί και όχι μόνο για τρεις ώρες την ημέρα γιατί ακόμα και οι ανθρωπιστικές οργανώσεις και τα Ηνωμένα Έθνη φτάνουν να είναι υποχρεωμένα να διακόψουν τις δραστηριότητες τους. Εάν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο έχουμε φτάσει πια σε ένα σημείο που δεν μπορούμε να δεχθούμε με κανέναν τρόπο. Η τρίτη αξίωση είναι η εντατικοποίηση της ειρηνευτικής διαδικασίας. Η μόνη βάση μπορεί να είναι η μόνιμη και διαρκής λύση δύο κρατών, Παλαιστίνης και Ισραήλ, ως κυριάρχων κρατών μέσα σε ασφαλή σύνορα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με τα συμβαλόμενα μέρη της τετραμερούς, μαζί με τις ε, αραβικές χώρες, πρέπει να συμβάλλει σε μια επιτυχή προσπάθεια λύσης, που αυτή όμως προϋποθέτει μια συμφιλίωση πρωτίστως και κυρίως συμφιλίωση μεταξύ των ομάδων των Παλαιστινίων. Οφείλουμε σήμερα να αναρωτηθούμε σχετικά με την μεθοδολογία την οποία χρησιμοποίησαμε μέχρι τώρα σε μια λεγόμενη ειρνευτική διαδικασία, παρόλες τις γνωστές δυσχέρειες, παρόλο, παρόλες τις ελάχιστες επιτυχίες, μέχρι που λίγο εβδομάδων μπορούσαμε να θεωρούμε ότι βρισκόμασταν μέσα σε μια λογική των διαπραγματευτικών διαδικασιών. Ολόκληρη η διεθνής κοινότητα και πρωτίστως η Ευρωπαϊκή Ένωση παρακολουθούσαμε και συνοδεύαμε και υποστηρίζαμε χρηματοδοτικά την προσπάθεια αυτή, διασφαλίζοντας τις συνθήκες πλαίσια για την ίδρυση Παλαιστινιακού κράτους. Αυτή η δέσμευση ήταν επαρκής, οφείλουμε να το αναρωτηθούμε. Στο μεταξύ η λογική αυτή έχει αντικατασταθεί από μια κλιμάκωση της βίας και αναγκάζει όλους να σκέπτονται βραχυπρόθεσμα. Αυτό που χρειαζόμαστε λοιπόν πρωτίστως είναι όντως μια εκεχηρία, μια άμεση ανακοχή και αποχώρηση των Ισραηλινών στρατευμάτων όπως ζήτησε και στο ψήφισμά του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Τα διδάγματα των τελευταίων δεκαετιών μας διδάσκουν ότι η ειρήνη δεν μπορεί να προκύψει στη Μέση Ανατολή μόνο μέσα από τις ίδιες τις προσπάθειες της περιοχής αυτής. Θα χρειαστεί υποστήριξη από όλες τις πλευρές. Γι' αυτό και πρέπει η διεθνής κοινότητα να είναι έτοιμη να υποστηρίξει και να προωθήσει την ειρήνη στη Μέση Ανατολή με κάθε δυνατό μέσο, ώστε να μπορέσουν να ξεπεραστούν οι πικρές εμπειρίες των τελευταίων δεκαετιών. Διεθνείς δυνάμεις μπορούν και πρέπει να συμβάλλουν στην διασφάλιση της ανακοχής αυτής. Το Γάλλο-Αιγυπτιακό σχέδιο για την ίδρυση ενός διεθνούς μηχανισμού για την προστασία και φύλαξη των συνόρων της Γάζας πρέπει να επιτύχει. Και αυτό βεβαίως πρέπει κυρίως να έχει ως στόχο τον αποκλεισμό της λαθρέας εισαγωγής όπλων στη λωρίδα της Γάζας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δηλώσει ότι είναι διατεθειμένη να αναλάβει δράση προς την κατεύθυνση αυτή. Η διεθνής κοινότητα δεν μπορεί όμως να ζητήσει και να διασφαλίσει μοναχά βραχυπρόθεσμα την ανακοχή θα πρέπει να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη που είναι απαραίτητη για την επανέναρξη των, δια, ε, διαπραγματεύσεων για την ειρήνη. Και αυτό σημαίνει ότι με την ενδεχόμενη αποστολή δυνάμεων οι οποίες πρέπει να έχουν μια ισχυρή εντολή θα μπορέσει μόνο να εξασφαλιστεί μια βάση για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης. Δεν μας αρκούν οι δηλώσεις υπέρ της ειρήνης που έχουν ακουστεί τόσο συχνά στο παρελθόν. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι η διάθεση, η προθυμία, όχι μόνο να προωθήσουμε την ειρήνη, αλλά να την διασφαλίσουμε πριν κλιμακωθεί ακόμη περισσότερο η κατάσταση και επεκταθεί και σε άλλες χώρες. Υπενθυμίζω ότι το 2008 υπήρξε το Ευρωπαϊκό Έτος του Διαπολιτισμικού Διαλόγου. Υπενθυμίζω πόσο πολύ εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταβάλαμε προσπάθειες ώστε το έτος εκείνο, το 2008, να γίνει έτος ελπίδας και να δώσουμε πολιτικές κατευθύνσεις που να δείχνουν ότι αυτή η λεγόμενη σύγκρουση των πολιτισμών δεν είναι δά και κανένα φυσικός νόμος. Δείχνουν όμως τα γεγονότα στη Γάζα πόσο γρήγορα μπορούν να καταστραφούν οι καλές αυτές ιδέες που προωθούμε σιγά σιγά και πετραδάκι πετραδάκι. Ακόμα χειρότερα, η πραγματικότητα αυτή ρίχνει νερό στους μήλους των εξτρεμιστών και των φανατικών που δεν έχουν στόχο την ειρήνη αλλά την περαιτέρω κλιμάκωση των συγκρούσεων. Η βία οδηγεί στην βία. Αυτό οφείλουμε να το επαναλαμβάνουμε ώστε να το αντιληφθούν όλοι. Μόνο ο διάλογος και οι διαπραγματεύσεις μπορούν να αποτελέσουν διέξοδο από την κρίση. Διάλογος και διαπραγματεύσεις δεν μπορούν να είναι αυτό ο σκοπό. Πρέπει να έχουν ως απότερο στόχο οι άνθρωποι στο Ισραήλ και στην Παλαιστίνη να μπορούν να διαβιώσουν σε πραγματική ασφάλεια, σε ειρήνη και με σεβασμό τη αξιοπρέπεια τους. Σας ευχαριστώ κυρίε και κύριοι συνάδελφοι για την προσοχή σας. So, liebe Συνεχίζει ο πρόεδρος Πέτερινγκ. Τα πρακτικά της συνεδρίασης της 5 η 18 Δεκεμβρίου 2008 έχει διανεμηθεί, έχουν διανεμηθεί. Υπάρχουν σχόλια. Όχι. Θεωρώ λοιπόν ότι εγκρίνεται. Οι αρμόδιες ρουμανικές αρχές μου ανακοίνωσαν ότι οι βουλευτές